Καταρχήν, έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση, πολύ σημαντική για όλους σας. Παρακαλώ την προσοχή σας. Koleżanki i Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισάγουμε το Wi-Fi. Χάρη σε αυτό θα μπορείτε να αξιοποιείτε το διαδίκτυο και να έχετε πρόσβαση σε αυτό σε όλα τα κτίρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα smartphones, τα notebooks, οτιδήποτε. Το σήμα δεν ε, υπάρχει μόνο στους χώρους της Ολομέλειας και των Επιτροπών ή άλλων αιθουσών συνεδριάσεων, αλλά και στους ευρύτερους γενικότερους χώρους. Δηλαδή εννοώ οπουδήποτε βρίσκεστε στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Wi-Fi. Αυτό συνιστά μια τεράστια αλλαγή στην ε, διαχείριση του χρόνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με αυτή την ευκαιρία επιθυμώ να συγχαρώ την ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης Υψηλής Τεχνολογίας και τον κύριο Ράινερ Βίλαντερ που κάθεται δίπλα μου, ο οποίος με μεγάλη επιμέλεια έφερε εις πέρας αυτό το εγχείρημα. Η διαθεσιμότητα του Wi-Fi είναι μία από τις πολλές καινοτομίες μας φέτος και υπενθυμίζω ότι η διεύθυνση High και ο συνάδελφος αντιπρόεδρος μας διέθεσε ένα EP Directory, ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και το e-committee ε, ε, Europarl Mobile και το IPEX website. Όπως βλέπετε, έχουμε επιφέρει πολλές βελτιώσεις φέτος που διευκολύνουν το έργο μας. Πάλι λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους τους ε, συνεργάτες του Κοινοβουλίου από όλες τις υπηρεσίες την Γενική Διεύθυνση και τον συνάδελφο Βίλαντ. Κυρίες και